των γειτονικών χωρών. Συγγνώμη, Possiamo riprendere il dibattito. Λοιπόν, μπορούμε να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Και πρώτα θα ακούσουμε το Συμβούλιο, εξ ονόματος του οποίου θα μιλήσει ο Υπουργός Νικόλας Εσμιτ. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Voilà. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Αμέσως, αμέσως. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Τα αίτια των ροών ε, προσφύγων που φτάνουν σε ακτές της Ευρώπης ε, εντοπίζονται στις κρίσεις και τους πολέμους στη Συρία και το Ιράκ, αλλά και της κρίσης ε, που αντιμετωπίζει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το Αφγανιστάν και το κέρας της Αφρικής. Η απόφαση που έλαβαν οι αρχή και κυβερνήσεων στην άτυπη συνόδο της 23ης ε, Συμβουλίου επιβεβαιώνει την ε, δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια αντιμετώπιση ανθρωπιστική, εσωτερική και εξωτερική πτυχή αυτής της κρίσης. Πολύ συγκεκριμένα αποδεσμεύουμε τους απαραίτητους για την επαναχρηματοδότηση των ανθρωπιστικών δράσεων και οργανώσεων πόρους, συγκεκριμένα για την ύπατη αρμοστία και το επιστηστικό πρόγραμμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα ε, όποια ανάγκη πιστιστική των προσφύγων όσο δυνατόν πιο κοντά στη χώρα προελεύσεως και μιλούμε για Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ. Στη Συρία παραμένουμε ο κύριος χορηγός εν ώψη του ε, χωρίς πόλεμο πολέμου που γνωρίζει η χώρα αυτή. Ε, απευθυνόμαστε ως το δυνατόν σε καταπιστεύματα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε συγκεκριμένα δράσεις για να βοηθήσουμε σε κρίσιμα θέματα όπως είναι η εκπαίδευση, η απασχόληση των νέων τους πρόσφυγες και ε, το Ταμείο Μαντάντε, παραδείγμα, το οποίο έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα υποχρηματοδότηση, αλλά και το αντίστοιχο τη Αφρική, βρήκαν ανταπόκριση κοινή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του κρατών και κυβερνήσεων στο πρόβλημα τη χρηματοδότηση. Στο εξωτερικό σκέλο αυτά, στο εσωτερικό σκέλο, έχοντα ε, επίγνωση τη έκταση τη κρίση και τη ανάγκη να δοθεί γρήγορη απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων, ε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα ε, και κατά προτεραιότητα. Δύο συνεδριάσεις λοιπόν του Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών έλαβαν χώρα στις 14 και 22 αντίστοιχα Σεπτεμβρίου του 2015 πέραν των ήδη προγραμματι... Ε, συνεδριάσεων από την Προεδρία και προκειμένου να εξασφαλιστεί για ε, η συνέχεια των όσων είχε αποφασίσει για, τον, ε, για την μετανάστευση και σε σχέση με τα μέτρα και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ήδη το καλοκαίρι και την άνοιξη του Συμβούλιο και με τις νέες προτάσεις Επιτροπής του Σεπτεμβρίου. Στη συνεργασία με τους Υπουργούς ε, της Επασχόλησης, εχθές μόλις και στο πλαίσιο του γεύματος ε, των Υπουργών, ε, προέβημεν σε μια ανταλλαγή απόψεων για την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή συγκεκριμένα στα κράτη τα οποία υποδέχονται το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων αυτή τη στιγμή, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους, προκειμένου επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η παροχή μαθημάτων γλώσσας, ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση των παιδιών και ούτε καθεξής. Η Επίτροπος κυρία Τάισεν μας ε, παρουσίασε μια σειρά από σκέψεις σε σχέση με την αξιοποίηση πόρων προερχομένων αφενός με κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα αυτά και η Επίτροπος έχει την πρόθεση και στο πλαίσιο του ΕΠΣΚΟ να συνεχίσει την επεξεργασία του, του θέματος έτσι ώστε κατά τρόπον συνεκτικό και αλληλέγγυο να προσφέρει μια προσέγγιση για τις χώρες εκείνες οι οποίες υποδέχονται το μεγαλύτερο αριθμό των προσφύγων. Όλες αυτές οι προσπάθειες επέτρεψαν και οφείλουν να επιτρέψουν να φτάσουμε σε συγκεκριμένα και σημαντικά αποτελέσματα στις συντομότερες δυνατές προθεσμίες και κυρίως με την υιοθέτηση 14 Σεπτεμβρίου μιας απόφασης του Συμβουλίου που θεσπίζει προσωρινά μέτρα προστασίας, διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα που επιτρέπουν δηλαδή την επανεγκατάσταση μιας πρώτης ομάδας 40.000 προσφύγων η απόφαση δε της 22 Σεπτεμβρίου ε, με την οποία το Συμβούλιο Υιοθετεί μια δεύτερη απόφαση για επανεγκατάσταση 120.000 ε, ατόμων χρηζόντων διεθνού προστασία από την Ιταλία και την Ελλάδα ή από οποιοδήποτε άλλο κράτο θα είχε αντίστοιχη ανάγκη σημαίνουν και διαπιστώνουμε ικανοποίηση πως ε, έχουμε προχωρήσει τα, ε, πρώτα, τα κέντρα διαλογής hot spot έχουν ε, ήδη καταστεί λειτουργικά περιμένουμε πολύ σύντομα και τα επόμενα έχουν γίνει ήδη σημαντικές πρόοδοι από την Ιταλία και την Ελλάδα που παρουσιάστηκαν στο φόρουμ εμπειρογνωμόνων με την Επιτροπή και σε συνεργασία με την ΕΑΣΟ και βέβαια ε, με τη συνεργασία της Στρατηγικής Επιτροπής για το Άσυλο με τη συνεδρία της 5ης Οκτωβρίου κατά την οποία εξετέθηκαν οι πρακτικές πτυχές της επανα, επανεγκατάστασης λεπτομέρειές τους. Το Συμβούλιο χαίρεται για την ιδιαίτερα καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο για την εξέταση αυτών των αποφάσεων και την υλοποίησή τους. Αυτό αποδεικνύει βούληση για δράση και ουσιαστική προστασία και βοήθεια στους πρόσφυγες. Και ιδιαίτερα στα πιο εκτεθειμένα σε βοήθεια και υποστήριξη κράτη. Αυτά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια και υποστήριξη δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί, ξεκινώντας από τη Λιβύη, διασχίζουν την Νότια Μεσόγειο. Εδώ περιμένουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συνεργασία με τους εταίρους μας στη Συνόδου της Λαβαλέτα είτε πρόκειται για τη μετανάστευση, είτε πρόκειται για τους πρόσφυγες, είτε πρόκειται για την καταπολέμηση των λαθροδιακινητών, αλλά και στην επαναπροώθηση ως Προεδρία Πρόεδρε. Εμείς ενεργά δραστηριοποιούμεθα για να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη αλλά και τους κυρίους εταίρους ώστε να ενισχύσουμε τη συμβολή και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό ώστε να φτάσουμε στο ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ που θα υποστηρίξει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κρίση αυτή. Οι κάτω χώρες και το Βέλγιο προεξήγηλαν επιπλέον 48,5 εκατομμύρια η μία και 30 εκατομμύρια ευρώ η άλλη ε, για το ίδιο θέμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο μιλάει για 100 εκατομμύρια λίρες. Η Γαλλία και η Γερμανία ε, ανακοινώνουν ότι θα θέσουν επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ εκάστη. Οι προσπάθειες αυτές στις οποίες πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποστηριχθούν και από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Και εν προκειμένου χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι η Γερμανία προεδρεύουσα του G7, της ομάδας των 7, οργανώνει την υπουργική διάσκεψη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών με ένα λεγόμενο outreach event ε, που επέτρεψε τη συλλογή επιπλέον 8 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει προτάσεις για προσαρμογή των δημοσιονομικών προβλέψεων και του προϋπολογισμού και εμείς ως Προεδρία είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε την ε, προσέγγιση αυτή στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αλλά βεβαίως χρειαζόμαστε και την ενεργό υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε γρήγορα σε μια απόφαση για τις αναγκαίες δημοσιονομικές προσαρμογές. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε προκειμένου να στηριχθούμε στην υποστήριξη σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Merci. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Σμιτ, ευχαριστούμε την Προεδρία του Λουξεμβούργου να δώσω αυτή αμέσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Τίμερμαντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα δοκιμαζόμαστε όλοι. Αντιμετωπίζουμε σαφώς τη μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρώπης εδώ και μια γενιά. Αυτό που δοκιμάζεται λοιπόν είναι η δυνατότητά μα να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό που δοκιμάζεται σήμερα είναι η δυνατότητά μα να κατανοήσουμε ότι λύσει θα υπάρξουν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που δοκιμάζεται είναι ακριβώ ο ίδιο ο ιστό τη κατασκευή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που δοκιμάζεται είναι οι θεμαλιώδει μα αξίε. Αυτέ που μοιραζόμαστε και πολλά υπόθηκαν ήδη το πρωί που το καταμαρτυρούν. Πρέπει να σημειώσω ότι όταν λένε κάποιοι, προσπαθούν να επιχειρηματολογήσουν ότι όσοι φτάνουν σήμερα στην Ευρώπη, κατά πλειοψηφία, είναι άνθρωποι που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον και όχι πρόσφυγες, αυτό είναι τελείως ε, μη αποδείξιμο. Δεν υπάρχει κανένα επιστημονικό στοιχείο. Ε, πολλοί εδώ στο σώμα σας το λένε και ε, αυτό μου δίνει κάποια ελπίδα τουλάχιστον ότι δεν θέλουν να φανεί ότι δεν κάνουν κάτι για τους αληθινούς πρόσφυγες. Δεν μπορείτε λοιπόν να απορρίπτετε ό,τι και να κάνουμε. Ε, κάποια πράγματα έχουν, όσο σήμερα μάλλον, έχουν να κάνουν με κατά πλειοψηφία πρόσφυγες. Αυτοί λοιπόν που επικρίνουν θα καταλάβουν πώς απατηλάνε τα επιχειρήματά τους και ότι μόνο ευρωπαϊκές λύσεις μπορούν να υπάρξουν εδώ. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από αυτό το γεγονός. Επίσης, υπόθηκε από εδώ και έτσι φαίνεται ότι η διαφωνία είναι ο τρόπο να έχει ένα επιχείρημα. Πηγαίνετε να του μιλήσετε στου καταβλισμού. Αυτό μου φωνάξατε. Μα αυτό και έκανα. Αυτό και έκανα. Αλλά προφανώ εσεί ακούτε αυτά που θέλετε όταν του μιλάτε στου καταβλισμού. Έτσι δεν είναι. Και ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτή τη φάση ο φόβο, ο φόβος είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για την ευρωπαϊκή κοινωνία, ένα σημαντικό παράγοντα. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε φοβούνται φοβούνται και ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό του φόβου. Όταν φοβάται κανείς πηγαίνει και ψάχνει στοιχεία για να βασίσει το φόβο του. Ε, δεν δέχεται αποδείξεις ότι ο φόβος είναι αβάσιμος ωστόσο, οπότε η ε, υπεύθυνη πολιτική στάση σε τέτοιες καταστάσεις είναι να μην τροφοδοτεί κανείς το φόβο να μην δημιουργεί στερεότυπα, να μην ομαδοποιεί και κατηγοριοποιεί τον κόσμο, αλλά να προτείνει λύσεις, λύσεις σε ένα πρόβλημα, αντί απλώς να διωγγώνει τους φόβους του κόσμου με την ελπίδα ότι θα πάρει περισσότερες ψήφους στις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η στιγμή που οι πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη ε, δέχονται την πρόκληση να δουν αν είναι ακόμη ακέραιοι ή αν θα επιλέξουν την πιο εύκολη λύση, την εύκολη διέξοδο, να τροφοδοτούν τους φόβους για να ενισχύσουν την πολιτική τους θέση. Ελπίζω ότι θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι σε αυτή την κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέδειξε υπευθυνότητα την περασμένη εβδομάδα, ξεκινώντα και ανοίγοντα το δρόμο για αποφάσει που τώρα μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται. Πολύ σύντομα να σα τι αναφέρω αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα να ενισχύσουν τα εξωτερικά σύνορα με αύξηση των οικονομικών κονδυλίων και των ανθρώπινων πόρων για του οργανισμού μα, τη Frontex, την ISO και την ε, Europol. Ε, αυξήθηκαν οι χρηματοδοτήσει για το ιστορικό πρόγραμμα τη ασφάλεια με 100 εκατομμύρια κατεπίγουσα ανάγκε για τα πλέον πληγέντα κράτη-μέλη. Ε, Επιπροσθέτω από τα 73 εκατομμύρια που ήδη έχουν δαπανηθεί. Πολλά από τα κονδύλια αυτά θα καλύψουν ανθρωπιστικέ ανάγκε προκειμένου να υπάρξει απαραίτητη στέγαση, η υγειονομική πρόνοια και οι άλλε βασικέ ανάγκε των νεοδικτέτων πρέπει να καλυφθούν. Επίση, επιταχύναμε τον επαναπατρισμό των ε, προσφύγων μα ε, με ομάδε βοήθεια και στήριξη στα λεγόμενα hot spot των ε, κρατών μελών, με την καταγραφή των αποτελεσμάτων των προσφύγων. Κάναμε διάκριση μεταξύ όσων έχουν δικαίωμα στο άσυλο και όσων όχι. Επίση, άρχισαν να εφαρμόζονται οι ισχύοντε κανόνε του Σέγγεν και του Δουβλίνου με περισσότερη προσοχή. Κινητοποιήθηκε η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για να συνδυαστεί με τι εθνικέ συνεισφορέ και ένα δι ευρώ για το επιστημιστικό πρόγραμμα ασφάλεια του ΙΕ, τη ΕΠΑ τη δηλαδή, αλλά και άλλα ειδικότερα προγράμματα για να καλυφθούν ειδικέ ανάγκε των προσφύγων στην περιοχή. Να στηρίξουμε την ε, Τουρκία, το Λίβανο και την Ιορδανία να αντιμετωπίσουν την κρίση με το ειδικό ταμείο για τη Συρία και με τα κατεπήγοντα μέτρα για την Αφρική αλλά και όσα αποφασίστη, θα αποφασιστούν στην ερχόμενη σύνοδο στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Είναι σημαντικές αποφάσεις. Ας τις υλοποιήσουμε επιτέλους. Εάν τις υλοποιήσουμε, το θέμα δεν θα είναι ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι όπως και σε άλλους τομείς, αυτό που μας λείπει είναι η αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας ε, το πρόβλημα. Όπως είπε και η Άγγελα Μέρκελ, μπορούμε. Απλώς πρέπει να μας απασχολήσει αυτό που θα έλεγα και σε αυτόν τον τομέα ότι υπάρχει περισσότερο ρίσκο. Πρέπει τα, τα κάτι μέλη να επιτεθούν, τα άλλα κάτι μέλη ότι μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλοι θα δραματίσουν το ρόλο τους και όλοι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και το έλεγχο στα εξωτερικά μας σύνορα. Όσοι φτάνουν στην επικρατειά μας θα πρέπει να ε, περνούν από έλεγχο δεκτυλικών αποτυπωμάτων. Όλοι θα πρέπει να επομιστούμε την ευθύνη που αυτή τη στιγμή επιβαρύνει μόνο μερικά κάτι μέλη. Αυτό είναι το θέμα εδώ λοιπόν κάνουμε όσα συμφωνήσαμε και η αυτοπεποίθησή μα όχι μόνο θα ενισχυθεί, αλλά και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα. Όπω είπα προηγουμένω και νομίζω ότι αληθεύει από πολλέ διαφορετικέ σκοπίε, Ο χειμώνα καταφτάνει. Μίλησα με τον Επίτροπο Κουτιέρη για του μετανάστε χθε και μου είπε ότι ξέρουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε από τις ε, μετρολογικές συνθήκες τους καταβλισμούς των προσφύγων. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τα κύματα ανθρώπων που θα βρίσκονται σε ε, διέλευση. Εφόσον κανείς ε, κινείται γρήγορα και άτακτα, είναι δύσκολο να προστατευτεί από τις σημερινές συνθήκες. Χθε οι συνομιλητέ μα καλωσόρισαν τα βήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιήσει κονδύλια για το σκοπό αυτό και να αναφέρω μερικά 200 ε, εκατομμύρια προ το επιστημιστικό πρόγραμμα τη Ορμοστία και άλλα ειδικότερα προγράμματα, 300 εκατομμύρια ανθρωπιστική βοήθεια του χρόνου και όπω ξέρετε ζητήσαμε από τα κάτι μελη να ε, αναλάβουν αυτή την ευθύνη σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Αυτά θα φανεί πω τι κατεύθυνση θα πάρουν ε, στο επόμενο Συμβουλίο, στην επόμενη Σύνοδο και θα καταλάβουν όλοι. Πιστεύω ότι ένα δις ευρώ δεν είναι πολλά για την ανθρωπιστική βοήθεια. Από αυτή τη σκοπιά είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων και προς το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί για άλλη μια φορά έδωσε το παράδειγμα και επιτάχυνε την υλοποίηση του προπολογισμού το Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο ανέλαβε τις ευθύνες του με τρόπο αξιοθαύμαστο. Η Συρία ε, με το ένα δις που θα με το ειδικό, μέσω του ειδικού ταμείου είναι κάτι το αξιοθαύμαστο εφόσον ο χειμώνα έρχεται. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κατεπίγουσα σήμερα, αλλά σε ό,τι αφορά τη βοήθεια αυτή δεν είναι μόνο ο στόχο να βρούμε τη σωστή χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να βρούμε και του απαραίτητου μηχανισμού βοήθεια, ε, ώστε να κινητοποιήσουμε ό,τι στοιχεία διαθέτουμε και αυτό είναι προτεραιότητε ε, των επιτρόπων Χαν Αβραμόπουλου, Στυλιανίδη, Αντριουκάητη για τα θέματα υγεία των προσφύγων. Ε, Θα πρέπει λοιπόν όλα τα μέτρα να τα ε, υλοποιήσουμε και μάλιστα αμελητή, χωρί να χάνουμε χρόνο άμεσα. Χρειάζεται ένα ε, άλμα για την ε, βοήθεια που θα πρέπει να προσφερθεί στην Ελλάδα, κάτι που γίνεται λόγω των καθημερινών αναγκών που παρουσιάζονται εκεί. Ο πρόεδρο Γιούνκερ μίλησε για την ανάγκη συντονισμού ε, των πόρων τεχνική βοήθεια και συνδρομή προ την Ελλάδα. Χωρί όμω δυνατότητε υποδοχή, τίποτε δεν θα λειτουργήσει και όλοι θα συμφωνήσουμε με αυτά. Η Ελλάδα με ένα ειδικό πρόγραμμα από την ειδική αρμοστία θα ενισχυθεί προ αυτό. Ολοκληρώνεται τι ερχόμενε εβδομάδε και η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο σύστημα του Δουβλίνου. Να, πρέπει εδώ να χαιρετήσω την δέσμευση της ελληνικής ε, κυβέρνησης ε, να επιστρέψει στο σύστημα του Δουβλίνου. Δεν είναι όλα έτοιμα για το χειμώνα, μεν, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, έχει ε, εντοπίσει όλα τα μέτρα που χρειάζονται σε επίπεδο δράσης και προπολογισμού και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός των σύνορων μας. Τουρκία, όπω είπε ο πρόεδρο Γιούνκερ, είναι η χώρα με την οποία θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και θα ενημερωθείτε και το απόγευμα πιο συγκεκριμένα για το τι θα κάνουμε τι ερχόμενε εβδομάδε. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ενώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την ευρωπαϊκή κατάσταση και να κατανείμουμε τι ευθύνε μεταξύ των ε, ενδιαφερομένων χωρών, εδώ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το ευρύτερο πρόβλημα κατά γενεσιουργά αιτία του φαινομένου αυτού. Ε, κάποια τα γνωρίζετε. Θα σταματήσω σε όσα είπε ο πρόεδρο Γιούνκερ για αυτά σήμερα το πρωί. Οι πρόσφυγες που τρέχουν να διαφύγουν από τον πόλεμο και τι διώξει, που μπορούν να ρισκάρουν τα πάντα για μια ευκαιρία να ζήσουν αξιοπρεπώ, θα συνεχίσουν να διαφεύγουν. Δεν έχουν επιλογή και δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή ούτε εμεί παρά να του προσφέρουμε ασφαλεί συνθήκε, να του προστατεύσουμε και να του φερθούμε όπω του αρμόζει και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλε χώρε, εκεί όπου μπορεί να φτάνουν σε πρώτη φάση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα κλίμα κοινή εμπιστοσύνη στην ε, ε, αντιμετώπιση αυτού του κατεπήγοντο ανθρωπιστικού φαινομένου και μαζί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς. Περνάμε στη συζήτηση τώρα. Οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν στις 12.30. Έχουμε 40 ομιλητές όμως. 40. Γι' αυτό παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Βόζεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κύριε πρόεδρε η συζήτησή μας για το προσφυγικό αυτή την ώρα συνδυάζεται άμεσα με την προηγούμενη συζήτηση. πολύ σωστά αναφερθήκατε ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει το μαχαίρι και το σπαθί για τη λύση αυτού του προβλήματος. η λύση πρέπει να δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά η λύση είναι πρωτίστως και κυρίως πολιτική. το λέω γιατί αναφέρθηκε πριν ο πρόεδρος τούσκ για την αλληλεγγύη των κρατών μελών που πρέπει να επιδεικνύεται και ορθώς για την προστασία των συνόρων για τον αναγκαίο σεβασμό στους κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης. όμως το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αν δεν υπάρξει άμεσα συνεργασία με τις χώρες προέλευσης του προβλήματος. ξέρετε πολύ καλά ότι η ευρωπαϊκή ένωση ένωση έχει κυρίαρχο λόγο στα αίτια που προκάλεσαν αυτή την προσφυγική κρίση αλλά κυρίως και πρωτίστως μια συμφωνία μνημόνιο με τις χώρες διέλευσης των ανθρώπων αυτών και αναφέρομαι στην τουρκία γνωρίζετε πολύ καλά ότι χτες ο πρόεδρος ερντογάν μας άσκησε κριτική γιατί δεν μπορούμε στα εδάφη μας να δεχθούμε την ανθρωπιστική κρίση 250.000 ανθρώπων όταν εκείνος φιλοξενεί δύο εκατομμύρια ξεχνώντας προφανώς ότι για αυτό τον αριθμό των προσφύγων χρηματοδοτείται γερά και ξεχνώντας προφανώς ότι υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής με την ευρωπαϊκή ένωση από το 2011 και με την ελλάδα με το 2014 που δεν τηρούνται. με αυτό θέλω να πω ότι αν όλοι δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους η ευρωπαϊκή ένωση η ευρώπη τα κράτη μέλη δεν μπορούν να, να δώσουν τη λύση σε ένα πρόβλημα που πρωτίστως και κυρίως έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και την επιβίωσή του. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και κύριος που τηρήσατε το χρόνο σας, ο κύριος Φλέκενστάιν για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες, όχι μόνο στα δικά μας κράτη-μέλη, αλλά και καθοδόν στη Βαλκανική και στην Τουρκία. Και βεβαίως στην ίδια την περιοχή της κρίσης. Και βεβαίως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές που με μεγάλη αυταπάρνηση και μέχρι εξαντλήσεως ε, ε, βοηθούν ε, στην ίδια περιοχή, στη Συρία, στη Σερβία ή στο σταθμό του Μονάχου. Είναι σωστό αυτό που αποφάσισε το Συμβούλιο να προβούμε από κοινού σε ε, μεγαλύτερα βήματα και σε Πού θα βρισκόμασταν όμω σήμερα ή τι θα είχε γίνει εάν τα κράτη-μέλη είχαν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους, δεσμευσει που, είχαν αναλάβει προπολού. Πού ε, ε, έχει παραμείνει το 0,7% για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να επιταχύνουμε και τις πληρωμές και τη δράση μας οι πρόσφυγες που έχουν υποστεί τα πάνδυνα και έχουν πλέον κουραστεί θα πρέπει να αξίζουν τον κόπο. Ευχαριστώ. Η κυρία Στέβενς για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συνάδελφοι. Η Τουρκία παίρνει τώρα οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, υποδέχεται και να συνεχίζει να αγκιάται την υποδοχή των προσφύγων. Ξεχνάει όμως τι γίνεται στη Συρία. Πολύ συχνά παραμένουν σε καταβλισμούς οι φτωχοί εκείνοι που δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν τη μεταφορά τους στην Ευρώπη. Ε, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη. Καμιά φορά επίσης χρειάζονται και ιατρική βοήθεια ή παραϊατρική. Αυτή η ειδική προσοχή είναι κάτι που δεν υπάρχει στους καταβλισμούς Ας πούμε, παιδιά με αναπηρία δεν μπορούν να πάνε σε κανονικό σχολείο. Ε, τι γίνεται με τη νοηματική γλώσσα. Τι γίνεται με το, ε, τη διδακτική ύλη ε, σε μπράι. Χρειάζεται ειδική βοήθεια για τους ανθρώπους αυτούς με αναπηρίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ή γίνεται σε πάρα πολύ ελάχιστο βαθμό. Διαπίστωσα όταν πήγα στον καταβλισμό Ζαατάρη στην Ιορδανία ότι υπάρχουν μεγάλε ανάγκε. Φέτος το Μάιο έγινε αυτό. Θα πρέπει τα μέσα αυτά να τα χρησιμοποιούμε με έξυπνο τρόπο και αποτελεσματικό. Και είναι σχετικά λίγα τα χρήματα που χρειάζεται και θα υπάρξει τεράστιο αντίκτυπο και βελτίωση τη ζωή των ανθρώπων αυτών στου καταβλισμούς. Ευχαριστώ. Κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την ευγνωμοσύνη μου προς τη Τουρκία, την Ιορδανία και το Λίβανο που μέχρι στιγμής έχουν υποδεχτεί 3 με 4 εκατομμύρια από τα 10 εκατομμύρια σύρων προσφύγων. Ενώ εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 28 μοντέρνες χώρες μας έχουμε μέχρι στιγμής ε, ε, υποδεχθεί περίπου 500.000. Είμαστε ε, η πιο πλούσια ήπειρος του κόσμου και αυτή είναι η συνεισφορά μας. Τώρα, τι γίνεται σε μερικά κράτη-μέλη. Ουγγαρία και τα δακτυλοδεικνύω. Τι συνάντησαν οι πρόσφυγες, σειρματοπλέγματα, φράχτες, ε, πυροβολισμούς, ε, δακρυγόνα. Χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνες βάρος των προσφύγων στην Ουγγαρία. Και επιπλέον η σημερινή εθνική νομοθεσία αναγνωρίζει και ε, μεριμνά ώστε οι Ούγγροι πολίτες που έδειξαν ελληνική και ανθρωπισμό και περιέθαλψαν στους, στα σπίτια τους ε, τους πρόσφυγες ε, διατρέχουν το κίνδυνο φυλάξη μέχρι και τριών ετών. Και μάλιστα οι γείτονές τους μπορούν να τους καταγγείλουν, ε, να, καταγγείλουν τους συνανθρώπους τους για, για, για, τον ανθρωπισμό και την ελληνική που έδειξαν. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε κύριε Πρόεδρε, αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε. Πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τέτοιου είδου νομοθεσία σε ένα κράτο και είναι πραγματικά επονίδιστο, επέσχυτο που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε τόσα περισσότερα πράγματα και τόσο καλύτερα, γιατί ο κόσμο μα κοιτάει, έχει στραμμένα τα μάτια του σε εμά. Ε, στα Ηνωμένα Έθνη, δυστυχώς ε, ο Όρμπαν στην ομιλία του ε, συγκέντρωσε την προσοχή στην Ευρώπη και σε αυτή την κατάσταση. Αν αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει στο μέλλον. Ο κύριος Χουαρίστη δεν είναι παρόν, η κυρία Σαρτζαντίνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους πρόσφυγες ε, λέει πολλά για τις αξίες, για την κοινωνία μας και για τις αρχές μας. Έχω μεγάλο θαυμασμό για εκείνους που μέρα νύχτα προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται σε μεγάλους αριθμούς και να τους ε, υποδεχτούν με τρόπο ασφαλή, σχολεία και αλλού. Αλλά πραγματικά εξοργίζομαι όταν βλέπω δακρυγόνα και ε, καθατό σειρματόπλεγμα σε κάποιες χώρες και τους πετάνε σάντουιτς πάνω από το φράχτη και τα σηματοπλέγματα. Έτσι βοηθάμε τους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε αυτά να τα αφήνουμε ατιμόρυτα, ε, διότι ε, θα επικρατήσει το χάος. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ε, να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ε, στην ε, Ουγγαρία της συμπεριφορά ε, του κυρίου Όρμπαν. Αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες συστηματικά εδώ πέρα αποκρούονται. Χτες το βράδυ από τους σοσιαλδημοκράτε. Μα αν δεν φορόμαστε πολιτισμένα ένα στον άλλον, πώς θα φερθούμε πολιτισμένα στους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. There is a blue card for you. θέλει να σας υποβάλει ερώτηση με μπλε κάρτα, κύριε Σαχερτίνη. Τη δέχεστε? Ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Εμείς τι περιμένουμε από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Να τηρούν τους ευρωπαϊκούς νόμους και να ε, φυλάσσουν τα σύνορα. Αυτό δεν είναι το σημαντικότερο θέμα και στην Ουγγαρία. Τα ουγγρικά σύνορα θα ε, έχουν περάσει από τη Σερβία και την Κροατία μέχρι σήμερα 300.000 άνθρωποι, η οποία Σερβία και ε, Κροατία ε, είναι ασφαλείς χώρες. Η Κροατία είναι μέλος, η Σερβία είναι ασφαλής χώρα. Γιατί πάνε στη Γερμανία, διότι είναι οικονομικοί μετανάστευση, τι πρόσφυγες. Έχετε το λόγο κυρία Σαρχεντίνη. Για να απαντήσετε. Κύριε, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι και επικεφαλής ε, της παρατήρησης των εκλογών στην Τανζανία και μου λέει ο κόσμος ότι παρατήρηση και ο έλεγχος δεν σημαίνει δράση. Αυτό που κάνει η ε, ε, Ουγγαρία δεν είναι παρατήρηση ούτε έλεγχος, είναι επαναπροώθηση και απόθηση pushback που απαγορεύεται. Φεράρα. Φεράρα. Grazie Presidente. Bene, να σας πω πως ε, αυτή τη στιγμή ακολουθούμε την ε, πορεία της ίσονος δυσκολίας. Ε, αυτή είναι η πηξίδα που μας καθοδηγεί. Τώρα, πρέπει να σας πω πως ήταν πολύ σωστές οι προσπάθειες που έχει με τις ποσοστώσεις και τους αριθμούς οποίους θα υποδεχθούμε. Νομίζω πως ε, με ένα πιλωτικό σχέδιο θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε και το Δουβλίνο έτσι ώστε να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό και να μην χρειάζεται κάθε φορά να περνάμε τέτοια μέτρα έκτακτα με μήνες αναμονής η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιο βαθμό αγνόησε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει πάντα ε, το προσφυγικό κείμενο, ε, κύμα. Είναι ε, παγκόσμιο πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχουν λύσεις πρέπει να δούμε όμως τι προκαλεί αυτά τα μαζικά κύματα. Είναι κάποιες ένοπλες συγκρούσεις, είναι η μάχη για την κατάκτηση φυσικών Ξέρετε πως το λόμπι των όπλων είναι πάρα πολύ δυνατό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρόσφατα ενέκρινε ένα ψησμά κατά ε, της πώληση όπλων μέσω παράνομων ε, οδών. έχουμε την επιχείρηση τρίτονας. Πιστεύετε πως επαρκεί για να μην χυθεί περισσότερο αίμα, για να μην ε, πεταχθούν τα λεφτά του Ευρωπαίου ε, φορολογούμενου. Εξ αντε προληπτικά ε, θα ε, δράει το Δουβλίνο ή εκ των υστέρων όταν έχουμε ήδη πνιγεί από το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φοντάνα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που με κλείσει περισσότερο στη συζήτηση παρά ε, τις ε, δικαιολογημένες διαμαρτυρίες κατά της Ουγγαρίας είναι ότι φαίνεται ότι παρα... ξεχνούμε το βασικό πρόβλημα που είναι η παρουσία του ίση στη Συρία. Δεν ξέρω τι επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ενώ μη ευρωπαϊκέ χώρε επεμβαίνουν στην κατάσταση, εμεί σιωπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε του Ήρου πρόσφυγε που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε τον πόλεμο. Και ελάχιστα κάνουμε για να το πραγματοποιήσουμε. Γιατί μιλούμε για φόβο, αλλά ε, εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχει φόβος και το γεγονό είναι ότι όλοι όσοι προκάλεσαν αυτό το κακό, όλοι όσοι προκάλεσαν αυτό το κύμα των προσφύγων, μένουν ατιμόρυτοι και δεν κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Και ο κύριος αυτούργός αυτής της καταστροφής είναι και υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Συναδίνος. Κύριος Συναδίνος. Πρόεδρε, πριν από ένα έτος ο Επίτροπος Αβραμόπουλος δήλωσε ότι δεν θα ξαναγίνουν τα κράτη της Ευρώπης κάστρα και αοριστολογούσε για πιθανή επανεξέταση των συνθηκών Σέγγεν και Δουβλίνου 2 ένα χρόνο μετά δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένο ή περήφανο με τα αποτελέσματα τη πολιτική του στο μεταναστευτικό. εκατοντάδε χιλιάδε λαθρομεταναστών έχουν κατακλείσει ευρωπαϊκέ χώρε οι εκατόμβε νεκρών στη μεσόγειο συνεχώ αυξάνονται τζιχαντιστέ επωφελούνται των μεταναστευτικών ροών για να διεισδύσουν στην ευρώπη. οι αρχέ των χωρών εισόδου αδυνατούν να ελέγξουν τι ορδέ των εισερχομένων πόσο μάλλον να προσφέρουν τα δέοντα στου πραγματικού πρόσφυγε και χώρε όπω η γερμανία η αυστρία και η σλοβενία επανέφεραν τους διασυνοριακούς ελέγχους ενώ άλλες χτίζουν φράκτες και χρησιμοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις τους στη μάχη για την επιβολή της τάξης και ασφάλειας. με ευχολόγια και επακτολούς χρημάτων δεν λύνεται το πρόβλημα. η ευρώπη οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να συνταχθεί στο πλευρό των χωρών που πολεμούν το ισλαμικό κράτος. πρέπει να εξαναγκάσει την τουρκία να πάψει να εκμεταλλεύεται τους λαθρομετανάστες και μάλιστα με χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένωση που διέρχονται από το έδαφος της και ως πρώτη χώρα εισόδου μουσουλμανική και γειτονική της συρίας να αναλάβει διεκπαιρέως των αιτήσεων ασύλου σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο και τον κανονισμό τη ΥΠΑΤΗΣ αρμοστία του οηε. ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς χαίρομαι που τα κράτη-μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα επιτέλους προχωρούν σε συγκεκριμένα βήματα. Και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι Αυτά που λέμε για ένα δις, για υποστήριξη πηγόντος και της ε, Τουρκίας να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα βήματα. Να υπάρξει εγγύηση ότι τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν αυξημένα και ότι θα ε, γίνονται πραγματικές πληρωμές. Γιατί μέχρι τώρα ε, στο επιστημιστικό ταμείο και πρόγραμμα ε, δεν τηρούνται ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από τα κράτη-μέλη. Ε, είναι πραγματικά εγκληματική αμέλεια που επικρατεί εκεί. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε και τα αίτια του πολέμου φυσικά και να μην τα αφήνουμε σε κάποιον που τελευταία στην Ουκρανία δεν διακρίθηκε πάρα πολύ για την φιλιρινική και τις καλές, ε, και τις καλές γειτονικές του σχέσεις. Επίσης, τι γίνεται με τα hot spots, με τα σημεία καταγραφής ε, και στη συζήτηση. Ε, βλέπω ότι η κυρία Σαρχεντίνη ε, προσπάθησε να επιτεθεί στους σοσιαλιστές και δημοκράτες και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διαφώνησε με αυτά που λένε οι πράσινοι και οι αριστεροί. Τα ίδια βλέπουμε στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Έχει σημασία λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέει ο πρόεδρος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τίμερμανς συγκεκριμένα βήματα και άλλη μεταχείριση για τους πρόσφυγες. Έτσι ώστε με νόμιμο τρόπο και συντεταγμένα να διαμορφώσουμε και τα περάσματα στα σύνορα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσο. Ο κύριος Αουρίστη που πριν έλειπε, αλλά δικαιολογημένα. Έχετε το λόγο. Άκουσα τα όσα είπε σήμερα το πρωί το Συμβούλιο και έχω την εντύπωση ότι απλώς θυματοποιηθήκαμε για να δικαιολογήσουμε το ότι κλείνουμε τα εξωτερικά σύνορα και με τον τρόπο αυτό λέμε ότι σεβόμαστε το Σέγγεν και φαίνεται πως η ασφάλεια είναι πιο σημαντική για μας από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάποια κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή αγοράζουν ε, και δέχονται τις ε, κραυγές της άκρας δεξιάς ε, για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πριν από ένα μήνα η κυρία Μογκερίνη είπε πως μία κρίση ε, μαζική προσφύγων που φτάνουν στην Ευρώπη μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Μα μιλάμε για το 1% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής, το 0,1% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πόσους ανοίγουμε τις πόρτες μας, σε 160.000 άτομα. Ξέρετε πως κάποια από τα δικά μας κράτη είναι οι βασικοί δωρητές στο Λίβανο, στην Ορδανία, στην ε, Τουρκία. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, αφήνοντας στην άκρη τις αυθύνες μας. Ας μην καλλιεργούμε το φόβο, το μίσος προς το διαφορετικό και να μην λέμε πως η ασφαλεία είναι πάντα υπέρ όλων, γιατί με τον τρόπο αυτό πάντα καταπνίγουμε στο τέλος τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα. Βάιντεν Χέλτσερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Με κάποιους συναδέλφους το Σαββατοκυριακό πήγα στο Λίβανο και την Ιορδανία και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ποια είναι η τεράστια επιβάρηση των κρατών αυτών. Ε, έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους και αναρωτηθήκαμε τι θα γίνει όταν εκραγεί όλο αυτό το σύστημα. Ήδη βλέπουμε ε, τι συμβαίνει με τις περικοπές της στήριξης. Τον Ιούνιο από 27 δολάρια το μήνα ε, μειώθηκαν στο μισό, 13 και μισό. Και αυτός ήταν ένας από τους λόγους για το μαζικό κύμα προσφύγων που ήρθαν στην Ευρώπη. Εγώ καλωσορίζω και χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου. Δυστυχώ φοβούμαι ότι έρχεται κατόπιν εορτή. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατεθούν αμελητή, ε, ουσιαστικά και πραγματικά και ε, κυρίως να είναι και περισσότερα. Αλλιώς θα έχουμε μαζικότατα και τεράστια προβλήματα. Χαλάχο. Κύριος Χαλάχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πατρίδα μου, η Φιλανδία, περιμένει γύρω στους 500.000 αιτήσεις ασύλου φέτος. 50, συγγνώμη, χιλιάδες. Δηλαδή, ε, δεκαπλάσιος αριθμός από τον συνήθι αιτήσιο αριθμό και οι περισσότεροι είναι νέοι από το Ιράκ, τη Σομαλία και την Υποσαχάρια Αφρική. Και έρχονται στη Φιλανθία γιατί οι λαθροδιακινητέ του υποσχέθηκαν ότι θα βρουν καλοπληρωμένη δουλειά, δωρεάν διαμέρισμα και ε, ζωή χαρισάμενη στην Ευρώπη. Ε, οπότε ε, τελικά καταλήγουν σε τρόγλες, σε καταβλισμούς, χωρίς φαγητό, γιατί δεν υπάρχουν ούτε δωρεάν διαμερίσματα, ούτε δουλειές έρχεται ο χειμώνα και θα έχουμε δεκάδε χιλιάδε απογοητευμένου ε, ε, και απεγνωσμένου, απόγνωση νεαρού στου δρόμου τη Φιλανδίας. Είναι επικίνδυνο και ανεύθυνο κύριε Πρόεδρε να επιτρέπουμε ε, τέτοια ανεξέλεγκτη μετανάστευση προ την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και ταχύτερα συστήματα επαναπατρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ. Εδώ και μήνους ολόκληρους συμφωνούμε όλοι ότι η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη είναι ιστορική σημασία. Σήμερα η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζει να διευρύνεται και ε, διαρωτόμαστε ποιε είναι οι αιτίε της, όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα, αλλά και στην καρδιά της ευρώπη Πριν λίγε μέρε με τη Μαριέλ Ντεσσαρνές πήγαμε στο διάδρομο αυτό των Βαλκανίων και πραγματικά εκεί είδαμε ζωφερές εικόνες που μας επανέφεραν στα μέσα του 20ου αιώνα και το, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είδαμε ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανήμπορους σε απόγνωση ε, που πήραν το δρόμο προς την Ευρώπη και περιμένουν από εμά μία απάντηση, κύριε Γιουνκέρ, άμεσης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και προς τα κράτη-μέλη και κυρίως στα κράτη που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης, στη Μακεδονία, τη Σερβία, για παράδειγμα. Και Φυσικά και βοήθεια στις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα. Ε, της Ευρώπης και θα πρέπει να συντονίσουμε το σύστημα των hot spots, ε, των κέντρων καταγραφής, όχι μόνο στα ε, χώρες με τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και στις κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να οργανώσουμε και να ελέγξουμε ταυτόχρονα αυτή την υποδοχή. Και αυτό χρειάζεται για να ελαφρύνουμε κάπως την πίεση από τα εξωτερικά σύνορα. Και μάλιστα θα πρέπει να γίνει επιτακτική αντιμετώπιση αυτού του θέματος, γιατί βρισκόμαστε στα πρόθυρα του χειμώνα. Παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο σας, μην ξεπερνάτε το χρόνο αγόρευσης, γιατί δεν μπορούμε να ε, καθυστερήσουμε τις ψηφοφόρειες ε, για μισή ώρα και παραπάνω. Γιατί ε, ο κάθε βουλευτής που δικαιούται λεπτό, αν μιλάει για 1,5 λεπτό, θα πρέπει να παρατείνουμε κατά μισό χρόνο το χρόνο της συζήτησης ε, και δεν τον έχουμε. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σμιτ, κύριε Τίμερμανς. Η συζήτηση αυτή αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ακούσαμε τίποτα γι' αυτό. Ακούσαμε κάποιες, κάποιους λογαριασμούς ε, και κάποια μέτρα, τίποτα για την κατάσταση των προσφύγων που είναι... Τι, ε, μιλάμε για μητρό και βλέπουμε να δίνουμε τροφή στους πρόσφυγες σαν να είναι άγρια θηρία. Ε, βλέπουμε να συνοστίζονται σε τρένα οι πρόσφυγες και να τους εγκαταλείπουν στη μέση του τίποτα. Βλέπουμε να συνοστίζονται σε καταβλισμούς προσφύγων με αναξεπρεπείς συνθήκες. Αυτή είναι η κατάσταση, η ανθρωπιστική κατάσταση χιλιάδων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συνθήκη που εγκρίνεται, η δική σας συνθήκη, λένε ότι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων βρίσκονται στις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν εφαρμόζεται η συνθήκη, εφαρμόζεται μόνο επιλεκτικά. Έχουμε τεράστια ανθρωπιστική κρίση ε, και τι θα κάνετε, τι θα, τι θα κάνετε με τον κύριο Όρμπαν, τι θα κάνετε στο φίλο σας, θα πρέπει να σεβαστεί τη συνθήκη ή αυτός ε, θα πρέπει να τύχει εξαίρεσης από τη συνθήκη. Ευχαριστώ. Micro, Με μικρόφωνο σας παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, Χαιρετίζω πολλά από τα στοιχεία των αποφάσεων του Άτυπου Συμβουλίου. Όμως πρέπει να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν, οι υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια στην ε, χερσαία οδό της μετανάστευσης θα έπρεπε να είχαν κληθεί τουλάχιστον στο άτυπο συμβούλιο. Οι πολιτικοί από το πρώην Σοβιετικό μπλόκο θα έπρεπε να γνωρίζουν περισσότερο τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της λήψης αποφάσεων υπέρ κάποιου ή μαζί με κάποιον ή και στη θέση κάποιου. Να σας υπενθυμίσω επίσης εσά στο Συμβούλιο πω αυτή η ειδική πλειοψηφία, η απόφαση που λήφθηκε με ειδική πλειοψηφία είναι θαραλέο μέτρο αν έχετε σκοπό να το πάτε μέχρι τέλου. Εάν δεν υπάρχει βούληση αυτή και δεν απαιτήσετε να επιβληθούν κυρώσεις στους όσους δεν συμμορφώνονται, απλώς μιλάμε για πολιτικό θέατρο και τίποτα παραπάνω. Κύριε Νάταλ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αμφισβητήσω το τίτλο της συζήτηση. Μιλάτε για κρίση προσφύγων. Γιατί, για να δακρύσουμε και για να εξυπηρετήσετε δικά σας πολιτικά συμφέροντα. Δεν είναι κρίση προσφύγων αυτή η κρίση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Είναι οικονομικών μεταναστών. Και αυτό δεν είναι απλώς η δική μου αξιολόγηση. Το είπε ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας. Είπε το 95% των ανθρώπων που έρχονται στην Ήπειρό μας δεν είναι πρόσφυγες είναι οικονομικοί μετανάστες. Όντως και η Eurostat, το δικό σας στατιστικό σώμα, είπε πως το 85% των ανθρώπων που έρχονται δεν προέρχονται από την Συρία, είναι από την Αλβανία, την Ιγυρία, το Πακιστάν, την Κάμπια. Τουλάχιστον ας μην προσβάλλουμε την ευφυία μας για να καλούμε αυτή την κρίση ε, με τον τρόπο αυτό. Μπορεί να μην το θεωρείτε πολιτικά ορθό, αλλά είναι κρίση οικονομικών μεταναστών, όχι προσφυγική κρίση. Κύριε Τίμερμανς, μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από φτωχές χώρες σε πιο πλούσιες χώρες. Και μεταξύ καταπατούν το διεθνές δίκαιο. Θα φαντάζονταν κανείς πως αυτό θα μας απασχολούσε. Όχι. Το μόνο που κάνουμε είναι να τους εθαρρύνουμε. Και υπάρχει βέβαια και η πτυχή της ασφάλειας σε τούτη εδώ τη φαρσοκομωδία. Μας είπε το ISIS πως θα πλημμυρίσουν την Ήπειρό μας με τους ε, ρηματικούς Ισλαμιστές. Κάνουμε κάτι να το αποφύγουμε. Όχι, το αντίθετο. Εμείς διακινδυνεύουμε τις ζωές ανθρώπων εδώ, εδώ, σε αυτούς που κάθονται πάνω, στην αίθουσα. Γιατί, Γιατί δεν σταματάμε αυτά τα κύματα. Οι γερμανικές αρχές είπαν ένας από τους τρεις Σύριους οι αυτοαποκαλούμενοι Σύριους φτάνουν με πλαστά διαβατήρια που αγοράζει κανείς για 750 ευρώ στην τουρκική μαύρη αγορά. Ποιοι είναι αυτοί. Μία από τις βασικές αρχές, θεμελιώδεις αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Δηλαδή αφήνουμε να μπούμε και έχουμε ελεύθερη, ε, ελεύθερη διακίνηση της τζιχάντ. Και νομίζω ότι όλοι θα έχουμε ματωμένα χέρια στο μέλλον επειδή ακριβώ πήραμε αυτέ τι αποφάσει. Κύριε Νάταλ. Διαδικαστικό. Διαδικαστικό, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι όλοι είμαστε εκλεγμένοι ευρωβουλευτές σε καθολικές ευρωπαϊκές εκλογές. Κύριε Τίμερμανς, είστε μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχετε δικαίωμα να επεμβαίνετε. Διακόπτει ο πρόεδρος. Εμείς έχουμε εκλεγεί από τους πολίτες, εσείς όχι. Δεν ήταν καθόλου διαδικαστικό. Παρακαλώ, α σεβαστούμε τον εσωτερικό κανονισμό. Ισχύει για όλους. Είστε ευρωβουλευτή, εκλεγμένο, ε, γι' αυτό πρέπει να σεβαστείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει υποβληθεί ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Νάταλ. Ο κύριο Καν. Μισό λεπτό όμω, παρακαλώ. Αν μου άνοιξε για το μικρόφωνο. Η ερώτηση είναι ότι ε, το Λίβανο, ο Λίβανος, η Ορδανία, ε, το Ιράκ, η Σερβία έχουν δεχτεί πρόσφυγες ε, από το, που έφυγαν, ξέφυγαν από το ISIS. Και τι έγινε, τι κάνατε, τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για το, για, ε, μα ήταν από, την, ε, από μια ε, οικογένειες από την Τουρκία που ήταν εγκαταστημένοι εκεί για πολλά χρόνια και ο πατέρας πήγε στον Καναδά προσπαθώντας να κάνει μια δοντιατρική επέμβαση, μια δοντιατρική αγωγή. Εδώ έχουμε οικονομικούς μετανάστες που έχουν κατακλείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέι, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν κάνουν τίποτα για αυτούς. Τι κάνουν? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Σαουδική Αραβία ε, πρόσφε, ε, πρότεινε στη Γερμανία να, να, να, ε, να λάβει 200.000 ε, Wahhabi. Συγγνώμη, 200 ε, τζαμιά στη Γερμανία για Wahhabites. Κυρία Κουντρίτσκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε ότι οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις επανεκατάστασης προσφύγων δεν είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Ευτυχώς αρχίσαμε ε, να αντιμετωπίζουμε και τις ε, αιτίε του κακού και να προσπαθούμε να βρούμε τα μέτρα για να τις αντιμετωπίσουμε. Αποτελεσματική ε, ε υπεράσπιση των εξωτερικών και έλεγχο των εξωτερικών συνόρων στη Μάλτα, στην Ελλάδα, είναι ο καλύτερο τρόπο για να επιλύσουμε την κρίση. Και η σωστή λειτουργική εφαρμογή των hot spot επίση είναι σημαντικό θέμα. Και θα πρέπει κατεπηγόντω να οργανώσουμε αυτό το θέμα. Και θα πρέπει να δούμε Πώ θα εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των μεμονωμένων προσφύγων. Πώ οι χώρες που θα υποδεχτούν τους πρόσφυγες που θα επανακαταστατούν θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια τους, ενώ πολύ συχνά έχουμε εμπριστικέ, ξενοφοβικέ ρατσιστικέ δηλώσει, γιατί αυτή είναι η απειλή που δημιουργείται κατά των προσφύγων. Το νέο προσφυγικό πακέτο δεν αρκεί λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε αναδιοργάνωση της ε, προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλίσουμε πραγματικό και πλήρη έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη εκστρατεία ενημερωτική για να πείσουμε τις τοπικές ε, αρχές ότι η υποδοχή των προσφύγων δεν απειλεί την ασφάλεια των ε, τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να δείξουμε αλληλεγγύη και ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπου που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Ευχαριστώ. Thank you. Κυρία Μακάβαν, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για πρώτη φορά το κοινοβούλιο μας συζητεί αυτά τα πράγματα την εσωτερική και την εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης μαζί. Νομίζω αυτό έλειπε μέχρι τώρα, μια συνολική ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πριν από λίγες εβδομάδες πήγα στην Τουρκία με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης και είδαμε πόσο μικρή είναι η συνοχή της πολιτικής μας εκεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε με την Τουρκία, είναι σωστό αυτό. Χωρίς την Τουρκία δεν υπάρχει λύση για το πρόβλημα. Θα πρέπει όμως να συνεργαστούμε και με τους οργανισμούς του ΟΗΕ. Τι είδαμε, περικοπές ε, στους προπολογισμού τους από τα κράτη-μέλη και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και βεβαίως ε, στην Τουρκία είδαμε πρόσφυγες, παιδιά που έχουν ακροτηριαστεί και είναι πρόσφυγες οι άνθρωποι αυτοί και δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Ε, απελπίζονται, είναι σε απόγνωση οι άνθρωποι, γι' αυτό έρχονται εδώ, θέλουν εκπαίδευση, παιδεία για τα παιδιά του. Εκεί χρειάζονται τα χρήματα και μια ε, ε, νόμιμη οδός να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νόμιμο τρόπο απευθείας από τους καταβλισμούς και η ΜΚΟ να ε, υποστηρίζονται αυτές που μπορούν να φτάσουν στη Συρία. Η ανθρωπιστική βοήθεια επιγόντως χρειάζεται. Sorry, there is a, there is a... Συγγνώμη, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Απαντήσετε. Παρακαλώ. 30 δεύτερα έχετε το λόγο. Τι προτείνετε δηλαδή, ότι θα φτιάξουμε και αυτοκινητόδρομο για το Ισλαμικό κράτος να περνάει τράνζιτ στην Ευρώπη. Τι γελία πράγματα είναι αυτά. Πού θα πάει η Ευρώπη. Θα αλλοιώσετε την ίδια τη φύση ε, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι παραφροσύνη. Να σας πω εγώ τι ξέρω. Πο, 15 μήνες είπε ο Νάιτζελ Φαράζ στην Βρετανική κυρία γνώμη ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες και τώρα έχουμε ευκαιρία να τους υποστηρίξουμε και εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει σύρος πρόσφυγας. Αυτά είναι φτηνά εκλογικά κόλπα. Ε, τα είπε και ο κύριος Τίμερ μας προηγουμένως. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι μπλε κάρτες επιτρέπονται για την υποβολή ερωτήσεων ε, για διευκρινήσεις από τον προλαλήσαντα Ευρωβουλευτή. Οι μπλε κάρτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε για συμπληρωματικές δηλώσεις, ούτε για προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Παρακαλώ να τηρήσουμε τον εσωτερικό κανονισμό. Ο κύριος Κρασνοντέμψκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στους καταβλισμούς προσφύγων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τραγική, δραματική. Και εκεί θα πρέπει να δρομολογήσουμε το μεγαλύτερο τμήμα της ανθρωπιστικής μας βοήθειας. Επιτέλους το καταλάβαμε. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όχι τα συμπτώματα αλλά τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Και αυτό απαιτεί τελείως διαφορετική πολιτική. Εκεί ίσως χρειαστούν και στρατιωτικά μέσα. Και σίγουρα δεν θα λύσουμε το πρόβλημα αν ανοίξουμε τις πύλες και τα εξωτερικά σύνορα για όλους τους πρόσφυγες και τους παράτυπους μετανάστες γιατί ακόμη και οι Γερμανοί σήμερα ε, επανήλθαν στην πραγματικότητα και προσγειώθηκαν και είδαν ότι και οι δικές τους ε, δυνατότητες είναι περιορισμένες. Όχι, δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα ούτε να σώσουμε τον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι η ανθρωπιστική λύση δεν είναι η υποχρεωτική επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη σε διάφορες χώρες στις οποίες δεν θέλουν οι πρόσφυγες ε, να μεταναστεύσουν και ούτε καν οι τοπικοί πληθυσμοί θέλουν να τους υποδεχτούν. Ευχαριστώ. Κύριε Κρασνοντέμψκι, Υπάρχει μπλε κάρτα για σας. Θέλετε να απαντήσετε. Ο κύριος Έθωριτς. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από τα είπατε είναι πολύ λογικά. Θα συμφωνήσετε μαζί μου πως ένα από τα πιο αειδιαστικά πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις εικόνες από απελπένους ανθρώπους έτσι ώστε να λυγίσει η καρδιά των ε, τηλεοπτικών ακροτηρίων έτσι ώστε να κερδίσουν κάποιο